συνάδελφοι, ακολουθούν επεξηγήσεις ψήφου. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους που αποχωρούν να το πράττουν όσο γίνεται πιο αθόρυβα. Euh, Έχω λάβει έξι αιτήματα για επεξήγηση ψήφου. Euh, λοιπόν, αρχίζουμε. Από τη σύσταση της κυρίας Αγιούζο. Για ένα λεπτό, το λόγο ο κύριος Κάρθη. Παρακαλώ. Σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Ευχαριστώ. Η σύμβαση για το διεθνές εμπόριο και τα απειλούμενα είδη της άγριας χλωρίδας και πανίδας ε, είναι ένα πολύ σημαντικό ε, νομικό μέσο και είναι σημαντικό να είναι μέλος αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρωταρχικός στόχος της σύμβασης είναι να εξασφαλίσει ότι το διεθνές εμπόριο ειδών ε, άγριας χλωρίδας και πανίδας δεν θα απειλεί την επιβίωσή τους. Πρόκειται για εμπόριο που σχετίζεται με την εκμετάλλευση ορισμένων φυτών, ορισμένων ζώων, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τους πληθυσμούς και μάλιστα ορισμένα ήδη να τα απειλήσει άμεσα με εξαφάνιση. Το εμπόριο ε, άγριων ε, ζώων και άγριας χλωρίδας ε, απαιτεί την διεθνή συνεργασία για να αποφευχθεί η επερεκμετάλλευση, για την προστασία επίσης της βιοπικιλότητας απαιτείται αυτή η συνεργασία γιατί μπορεί να επηρεάσει και λαούς ε, και επιχειρήσεις, βιομηχανίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Το ΣΥΝΦΕΙΝ υποστηρίζει λοιπόν το ψήφισμα αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Κινίτσι και αυτή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Διεθνή Σύμβαση Τσίτες προστατεύει 135.000 πανίδας και χλωρίδας. Η ένταξη στη Σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα σημαντικό βήμα, όχι μόνο γιατί γινόμαστε μέλος της Σύμβασης και θα παίξουμε σημαντικότερο ρόλο, αλλά γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργήσει ως πρωτοπόρος στην διεθνή πολιτική της προσπάθειας για διάσωση της βιοπικιλότητας μιας και έχουμε την πιο προχωρημένη νομοθεσία. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ε, δολάρια ε, τον χρόνο, είναι ο κύκλος εργασιών. Φυσικά είμαστε ο πρώτος εισαγωγέας σε ερπετά τύπου βόα στον κόσμο και σε πάρα πολλά επίσης ελ, η σύνδεση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σύμβαση αυτή θα ευνοήσει την καταπολέμηση αυτού του είδους των φαινομένων και γι' αυτό υπερψηφίζω την πρόταση. Η κυρία Γκέρλινγκ για ένα λεπτό και παρακαλώ ε, όσοι είστε στους διαδρόμους να φύγετε από την αίθουσα. EU Ευχαριστώ. Υποστηρίζω την προσχώρηση της Ένωσης ε, σε αυτή τη σύμβαση ε, ΣΥΤΕΣ. Αφού έχουν υπογράψει βέβαια τα περισσότερα κράτη-μέλη, γιατί ε, θα έπρεπε να υπογράψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια προστέμενη αξία θα είχε αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μιλούν πάντοτε τα κράτη-μέλη της Ένωσης με μια φωνή, αλλά υιοθετούν τελείως διαφορετικές θέσεις, παρότι έχουν προσυπογράψει την ίδια σύμβαση. Άρα αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα πρώτον να διαπραγματευτούμε μια νέα θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έπειτα πιστεύω ότι θα μπορούμε με το βάρος που έχουμε αντιπροσωπεύοντας όλους τους πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να αγωνιστούμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, διότι το εμπόριο εξωτικών ειδών είναι το τρίτο ε, σε κλίμακα παράνομο εμπόριο μετά τη διακίνηση ανθρώπων. Κύριε Γιάννη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι σχεδόν συμφωνούμε ότι είναι καλό που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρεί και προσχώρησε μάλλον στις σάιτες. Βέβαια, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί γιατί άραγε τόσο αργά. Η απάντηση είναι ότι μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατό αυτό. Μόνο κράτη-μέλη μπορούσαν να είναι μέλη ε, και όχι ενώσεις. Από τι 21 Νοεμβρίου του 2013 υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα και χαίρομαι που αδράξαμε την ευκαιρία μαζί ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ρίξουμε όλο μας το βάρος στη ζυγαριά και ε, σωστά είπαν οι συνάδελφοι θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε τώρα αυτό το βάρος. Είναι καλό αυτό για τον απελούμενο ε, κόσμο των ζώων ε, είναι πάρα πολλά τα είδη που απειλούνται κάθε χρόνο και είναι και πολλές οι παράνομες εξαγωγές. Και ένα τελευταίο ε, νέο που είναι λιγότερο ευχάριστο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να πληρώνει τέλη ε, συνδρομή εκεί που όμως θα είναι υπέρ των κρατών μελών γιατί θα πληρώνουν λιγότερες εθνικές συνδρομές στα κράτη-μέλη οπότε βγαίνουν κερδισμένα. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Το λόγο έχει ο κύριος Κόρμπετ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ συμφωνώ με τους συναδέλφους ακριβώς για τους ίδιους λόγους και καλωσορίζω την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση, αλλά έχω και έναν επιπλέον λόγο. Στην ίδια μου τη χώρα υπάρχει ένα είδος το οποίο είναι απειλή και αυτό ονομάζονται φιλοευρωπαϊκοί συντηρητικοί. Ε, έχουν πάρα πολλούς κυνηγού στο ίδιο τους το κόμμα και φυσικούς εχθρούς και θα πρέπει να καταχωρηθούν ε, ως ε, απελούμενο είδος και να αξίζουν και να τους δοθεί ιδιαίτερη προστασία από όσους τους επιτίθενται στο ίδιο τους το κόμμα. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ο κύριος Χάναν τώρα, για ένα λεπτό. Trade is not... Ευχαριστώ. Το εμπόριο δεν είναι κατά ανάγκη εχθρός ε, της διατήρησης ειδών. Το να δίνουμε κίνητρα στον κόσμο να αντιμετωπίζουν όμως τη χλωρίδα και την πανίδα ε, ως ε, ένα κομμάτι ε, του πλούτου, του φυσικού πλούτου, βοηθάει. Είδαμε τι έγινε στην Κένια που απαγόρευσε το κυνήγι ελεφάντων, ενώ η Τζιμπάμπουε τους ε, θεώρησε κληρονομιά. Και ήταν τελείως διαφορετικές οι εξελίξεις. Στη μία χώρα, ο στην Κένια συγκεκριμένα, ε, ε, αυξήθηκε πάρα πολύ ο πληθυσμός, γιατί θεωρήθηκε πολύτιμο ένα πολύτιμο ζώο. Τα 28 κράτη-μέλη έχουν υπογράψει την ε, σύμβαση, αλλά το θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να εκμεταλλευτεί περισσότερο αυτό το ενιαίο που της δίνει ε, η οντότητά της και να μας εκπροσωπεί στις διεθνείς, στα διεθνή βήματα συζήτησης. Η κάθε χώρα μπορεί βέβαια να αποφασίζει κατά το δοκούν και με βάση τις δημοκρατικές της διαδικασίες. Αλλά καλό να έχουμε μια ενιαία εκπροσώπηση. Για να ολοκληρώσουμε, ο κύριος Ντεμές Μάκερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το λαθρεμπόριο που απειλεί ε, τα άγρια ζώα και φυτά ένα παγκόσμιο πρόβλημα, άρα χρειάζεται παγκόσμια αντιμετώπιση. Η Διεθνή Σύμβαση ΣΑΙΤΕΣ είναι το πιο σημαντικό εργαλείο που έχουμε σε αυτή την ε, καταπολέμηση. Για όχι μόνο για να επιζήσουν αυτά τα ίδια, αλλά πρόκειται και για την ασφάλεια τη δική μας και την ειρήνη. Όλο αυτό το εμπόριο ε, έχει φτάσει σε ένα, μια μπίζνα δισεκατομμυρίων και χρηματοδοτεί πολέμους και τρομοκρατία δημοκρατία. Το κόμμα μου, NVA, υποστηρίζει απολύτως την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σάιτες και την υπερψηφίσαμε. Ήταν μόνο παρατηρητή μέχρι τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μπορούσαν να υπογράφουν μόνο κράτη-μέλη. Ε, και έτσι αυξάνεται και η δύναμή μας και η νομική μας ισχύ χωρίς να θίγεται καθόλου το θέμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνονται εδώ λοιπόν οι επεξηγείς ψήφου. Διακόπτε τη συνεδρίαση μέχρι τις 3 η ώρα. Καλή σας όρεξη